πράγματα. Νομίζω ότι ε, όσον αφορά τους αίθουσες θα πρέπει να πούμε κάτι για αυτό το θέμα εδώ στην αίθουσα. Πρόεδρος, η μέση διάταξη περιλαμβάνει τις προσωπικές ερωτήσεις προς την Κομισιόν σε σχέση με τις βάσεις δεδομένων όσον αφορά αθνητικές και φιλικές βάσεις δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινάμε τη συζήτηση, δίνουμε το λόγο στους συντάκτες, ξεκινώντας με την κυρία Φλασικόβα Μπενόβα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Καλησπέρα συνάδελφε. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα ΜΜΕ, η Γαλλική Αστυνομία χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων που περιέχει, που περιέχει στοιχεία για τους δρομά. Διάφορες ΜΚΟ διαμαρτυρήθηκαν για τη δημιουργία αυτής της βάσης δεδομένων που αφορά εθνοτικά και φιλετικά στοιχεία και έκαναν εκκλήσει προς τις αρμόδιες γαλλικές αρχές, οι οποίες όμως αρνούνται την ύπαρξη μια τέτοια βάσης δεδομένων. Είχαμε την ανακοίνωση ότι τα δεδομένα για τους Ρωμά θα πρέπει να φυλαχθούν σε μια νέα βάση δεδομένων, η οποία θα βρίσκεται υπό δημιουργία. Και η Ολλανδία, αλλά και άλλες χώρες φαίνεται ότι έχουν παρόμοιες βάσεις δεδομένων. Το Συμβούλιο φαίνεται να έχει φιλόδοξου στόχου όσον αφορά τι εγκληματικέ ομάδε και πρέπει να έχουμε και εμεί στο Κοινοβούλιο εδώ και μια αντίστοιχη πρωτοβουλία. Οπότε να ρωτήσω την Επίτροπο τι θα κάνει η Επιτροπή σε σχέση με την ύπαρξη αυτών των βάσεων δεδομένων στη Γαλλία και θα ήθελα να επαληθεύσει το κατά πόσο ισχύουν αυτές οι πληροφορίες. Δεύτερον, θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο η Γαλλία παραβιάζοντας στην αρχή τη μη διάκριση, τι μέτρα θα λεφθούν κατά τη Γαλλίας, αλλά και σε άλλες χώρες μέλη σε σχέση με τη δημιουργία ή ύπαρξη αυτών των βάσεων δεδομένων που περιλαμβάνουν φιλοτικά και εθνοτικά στοιχεία. Η υπαρξη αυτων των βασεων δεδομενων που περιλαμβανουν φιλοτικα και εθνικα στοιχεια η κομισιον θα ξεκινήσει μια έρευνα για την ανέρευση αυτών των βάσεων δεδομένων και θα διερευνήσει την ε, νομιμότητά τους υπό το φως του νόμου της μη, της μη τι συμβαίνει και στις χώρες μέλη όσον αφορά τις διοικητικές διαδικασίες οι οποίες ε, δεν θα πρέπει να καταλήγουν σε εθνικές διακρίσεις, εθνικές και διακρίσει. διακρίσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος τον κύριο Φλότρο για μισή λεπτά. Κυρία Φλότρο, συγγνώμη. Καλησπέρα κυρία Ρέντινγκ. Σήμερα θα μάθατε ότι η Γαλλία απάντησε στην ε, κλίση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εφαρμόζοντας αυτά που προβλέπει η οδηγία για την ε, ελεύθερη κυκλοφορία. Όπως είπατε και εσείς, δεν ακυρώνονται, αλλά αυτή η διαδικασία παραβίασης έρεται προσωρινά. Εμεί λοιπόν αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα ω Κοινοβούλιο, θα πρέπει να ασκήσουμε τα δημοκρατικά μα δικαιώματα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και τι υποσχέσει οι οποίε είχαν δοθεί από τι γαλλικέ αρχέ για το θέμα αυτό. Όλοι θα θυμάστε όμω ότι είχαμε ερωτήσει τη Γαλλία σε σχέση με τα έγγραφα που θα πρέπει να ελέγχονται στα σύνορα, σε σχέση με τον μη ε, χαρακτήρα διάκρισης αυτών των εγγράφων. Και τέλος, μετά από την εμφάνιση στο τύπο και βλέπουμε ότι πάλι στο τύπο εμφανίζονται πληροφορίες σε σχέση με μια βάση δεδομένων, με φακέλους οι οποίοι περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία τα οποία αναφέρουν την ε, εθνική ή φιλετική προέλευση των ατόμων αυτών. Μήπως λοιπόν εδώ δεν θα πρέπει να είμαστε και τόσο σίγουροι για την αξιοπιστία των γαλλικών αρχών. Κυρία Ρέντινγκ, δεν θεωρείτε απαραίτητο σήμερα να συνεχίσουμε και να μας πείτε σήμερα ποια είναι η δική σας ανάλυση. Η ανάλυση που βασίζεται σε δεδομένα που έχετε και στοιχεία που έχετε ζητήσει όσον αφορά τη δυνατότητα διαδικασίας παραβίασης για διακρίσεις εκ μέρους της Γαλλίας, αλλά επίσης και διαδικασία παραβίασης όσον αφορά τον νόμο για προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Νομίζω ότι σήμερα οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα να προσδοκούν μια υπεύθυνη κομισιόν επιτυχή, η οποία όμως θα δείχνει την αποφασιστικότητά της και την αυστηρότητά της όσον αφορά τις δράσεις της προς τις γαλλικές αρχές. Όπως κάνατε εξάλλου προς τις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ένωσης που όπως γνωρίζουμε έχουν κακή συνήθειες όσον αφορά τους ε, Ρώμα. Και σε σχέση με τους ε, φακέλους, η Εθνική Επιτροπή της Γαλλίας για την Ελευθερία διαπίστωσε την ύπαρξη τεσσάρων παρανόμων μητρώων που έφτανε στο σημείο μάλιστα να καταχωρεί και τη συγκεκριμένη προέλευση των ε, τσιγκάνων, ήταν Μανού, ήταν Ρώμ κλπ. κλπ. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ πολύ να τηρήσετε τις προθεσμίες, τις προθεσμίες το παρεμβάσεων σας γιατί έχουμε καθυστέρηση. Ιντφέλτ, τρία λεπτά. Κύριε Επίτροπε, ξέρουμε ότι είστε ένα άτομο θαραλέο και δεν θα επαναχωρήσετε, αν δεν θα υποχωρήσετε μάλλον, ξέρουμε ότι θα πάτε κατευθείαν στο στόχο σας και ευχόμαστε να είστε εξίσου αποφασιστικοί και σε αυτή την υπόθεση. Είχαμε την ανακοίνωση της Κομισιόν για την εφαρμογή της χάρτας των βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Κομισιόν λοιπόν θα πρέπει να κάνει πλήρη χρήση των ομοδιοτήτων της ώστε οι χώρες μέλη να εφαρμόζουν σωστά την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να σέβονται και να τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διαφορετικά θα ξεκινήσει η διαδικασία παραβίασης. Στην περίπτωση λοιπόν της Γαλλίας διερωτώμε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαφείται αποκλειστικά στις δηλώσεις των εθνικών κυβνήσεων, όπως είπε προηγουμένως η κυρία Φλότρο είχαμε μια σειρά δηλώσεων οι οποίες φάνηκαν να είναι αναξιόπιστες γιατί λοιπόν η Κομισιόν όπως έχουμε ζητήσει παλαιότερα δεν ξεκινά τις δικές της έρευνες και ελέγχους ώστε να γίνει κάτι. Ξέρετε ότι στο Κοινοβούλιο υπάρχει πλειοψηφία υπέρ των πράξεών σα. Είμαστε λοιπόν μαζί σα, κυρία Ρέντινγκ. Τώρα για την κατάσταση στη Γαλλία αλλά και για την κατάσταση στην Ιταλία η οποία φαίνεται ότι είναι σοβαρότερη και για την κατάσταση στη χώρα μου θα ήθελα να μάθω καταρχήν μπορεί η ύπαρξη αυτών των βάσεων δεδομένων να επιβεβαιωθεί Έχουμε αποδείξεις ότι υπάρχουν αυτές οι βάσεις δεδομένων ή όχι. Έχουμε ένα κατάλογο για την περίπτωση των κάτω χωρών ξέρω ότι υπάρχει κατάλογος επειδή οι δήμοι και οι κοινότητες που συντάσσουν αυτέ τι βάσει δεδομένων είναι και περήφανε, γιατί νομίζουν ότι έκαναν και καλή δουλειά, ίσω να είχαν καλέ προθέσει. δεν ξέρω. Αν λοιπόν υπάρχουν αυτέ τι βάσει δεδομένων θα θεωρήσετε ότι αυτό είναι νόμιμο ή όχι. Αν είναι νόμιμο τότε χρειάζεται να συζητάμε. Αν δεν είναι νόμιμο τότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε δικασία παραβίαση, Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή δεν διστάζει σε άλλους τομείς και εσείς είχατε μια τολμηρή στάση ανυποχώρητη όταν ασχοληθήκατε με, τις, με την περιαγωγή στην Ευρώπη. Αν υπάρχουν λοιπόν καρτέλ που δρούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διστάζει καθόλου. Και εδώ λοιπόν θα έπρεπε να δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Επιτροπή κυρία Ρέντινγκ θα πρέπει να αποδείξει ότι συμμερίζεται τι κοινοτικέ ευρωπαϊκέ αξίε τη στιγμή που έχουμε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μα παρακολουθούν οι πολίτε και όπω κυρία Φλότρο θα ήθελα να σα ζητήσω να έρθετε στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών και να μα εξηγήσετε πώ έχει η κατάσταση και τι δράσει προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ ω ε, ευρωβουλευτή και ω Ευρωπαίο πολίτη, θα ήθελα να μάθω όλη την αλληλογραφία που έλαβε χώρα μεταξύ ε, Κομισιόν και Γαλλίας και με τις υπόλοιπε χώρες μέλη επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δυόμιση λεπτά, Ernst. Κυρία κυρίες και κύριοι, θέτω το ερώτημα απλά. Τι γίνεται με την ίση μεταχείριση και μία αρνητική μεταχείριση των Ρωμά των Συγκάνων στην Ευρώπη. Όταν ακούμε τώρα ότι υπάρχουν τράπεζες δεδομένων και πιστεύω ότι απαγορεύονται τέτοιου είδους τράπεζες δεδομένων όταν έχουν την εθνοτική πτυχή που καλύπτουν και χρησιμοποιούνται από την γαλλική χωροφυλακή αστυνομικέ αρχέ για του τσιγκάνου. Και όταν μα λένε ότι γίνεται αυτό, λέει προφυλα... προφυλακτικά, προληπτικά. Ε, τότε έχει ξεχυλήσει το ποτήρι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και όταν συλλέγονται τέτοιου είδου στοιχεία για την εθνοτική προέλευση πολιτών, αυτό απαγορεύεται κάθετα και ρητά. Υπάρχει πολύ μεγάλο κίνδυνο αρνητική διακριτική μεταχείριση, μεροληψία και μόνο υπό πάρα πολύ αυστηρού όρου που δεν θα ε, ενέχουν μεροληψία, μεροληπτική αντιμετώπιση μπορούν ίσως να χρησιμοποιούν κάποιες τράπεζες δεδομένων. Εθνοτικές τράπεζες δεδομένων ως κυρώσεις και για προληπτικούς λέει σκοπούς είναι κάτι το οποίο παραβιάζει την νομοθεσία και είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται. Αναμένουμε και προσδοκούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε είδους εθνοτικών τέτοιων στοιχείων και φιλετικών στοιχείων ως στη συλλογή του και αποθήκευσή τους να την απαγορεύσει. Να πάψουν να υπάρχουν τέτοιε τράπεζε δεδομένων. Ειλικρινά σα λέω, διαρωτώ με όλο και περισσότερο. Λέμε, συζητάμε, λόγια, λόγια και πραγματικά έχει ξεπεράσει πια κάθε όριο αυτό. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την βελτίωση της κατάσταση των Ρωμά. Τι γίνεται πρακτικά χειροπιαστά πέρα από λόγια, λόγια, λόγια και να δούμε την συλλογή στοιχείων σε τράπεζε δεδομένων, ε τότε τι διαπιστώνουμε, ότι είναι ξυλαστήρια θύματα οι τσιγκάνοι και λαμβάνονται μέτρα απέλασή του σε πολλά κράτη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, απελάβνονται στο, κοσυφε, στο Επί μήνε παραβιάζει η Γαλλία ε, ε, ευρωπαϊκές και ευρωπαϊκή νομοθεσία και είναι αυτάρεσκοι και ικανοποιημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση με την υπόσχεση λέει της, Ευρω... γαλλικής μέχρι την αρχή του 2011 την νομική βάση για την υλοποίηση λέει, της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων να την διασφαλίσει. Αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι να πούμε τότε να σταματήσουν οι απελάσεις των Ρωμά, των συγκάνων από πλευράς Γαλλίας. Και εκείνοι οι ε, Ρωμά που έχουν απελαθεί θα πρέπει με ε, διευκολύνσεις και με συνοπτικές διαδικασίες να επιτραπεί να επιστρέψουν στη Γαλλία. Ποιες πληροφορίες έχετε λοιπόν εσείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποιες πρωτοβουλίες και διαβήματα κάνετε όταν γνωρίζετε ότι υπάρχουν τέτοιες ε, τράπεζες δεδομένων. Θα έπρεπε ε, για παραβίαση των ευρωπαϊκών συνθήκων να ασκήσετε προσφυγή βάρο τη Γαλλία Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Επίτροπο έχει το λόγο. Νομίζω ότι τόσο αργά που δουλεύουμε είναι κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συζητάμε ένα τόσο σημαντικό θέμα το οποίο θα έπρεπε να συζητάμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και όχι τα μεσάνυχτα όπου οι κανονικοί άνθρωποι θα έπρεπε να πηγαίνουν για ύπνο τώρα. Πέραν αυτού, έχουν προηγηθεί πάρα πολλές συζητήσεις, έχουν προηγηθεί πολλά σκάνδαλα και πολλές ενέργειες τις τελευταίες εβδομάδες. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δει το τι ακριβώς συνέβη στη Γαλλία και το τι αντιδράσεις υπήρξαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν κάτι το οποίο ήταν μια ιστορική στιγμή θα έλεγα. Μέχρι τώρα ποτέ στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπήρξε μια δικαστική διαδικασία η οποία να ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ξεκινήσαμε τέτοιες διαδικασίες επί παραβιάση, επί παραλήψη για τα οικονομικά ή για άλλους λόγους, αλλά η μοναδική περίπτωση ε, στην οποία βασιστήκαμε για την προσφυγή αυτή στη Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι αυτή. Είπαμε αρκετά σαν Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Και ομόφωνα λοιπόν 27 επίτροποι στις 29 Σεπτεμβρίου αποφάσισαν να ξεκινήσει η διαδικασία εις βάρος της Γαλλίας επί τη βάση της μη εφαρμογής από πλευράς της αυτών των δικαιωμάτων του ανθρώπου, των δικαιωμάτων του ατόμου, του μεμονωμένου πολίτη. Δεν χρειάζεται να σας επαναλάβω όλες τις διαδικασίες οι οποίες ακολουθήθηκαν από τότε. Είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ομόφωνα επαναλαμβάνω, ότι θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες αυτές επί παραβιάση και θα θέσουμε μια τερματική προθεσμία χρονική στη Γαλλία και αν δεν έχει αντιδράσει θετικά η Γαλλία μέχρι τις 15 Οκτωβρίου τότε η δικαστική αυτή διαδικασία θα ξεκινήσει. Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε. Προηγείται μια περίοδος προειδοποίησης. Λοιπόν, η Γαλλία έδωσε μια απάντηση είναι η πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, μοναδική φορά σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίσαμε τέτοιου είδους προβλήματα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το συμβάν αυτό είναι ίσως μια κεντρική στιγμή για την Ευρώπη των πολιτών. Αλλά αυτό ας το εξετάσουν οι ιστορικοί. Η διαδικασία έχει τώρα ξεκινήσει, βρισκόμαστε στη μέση της και μπορεί ο καθένας να έχει τις γνώμες τους. Τι λέει η Γαλλία, τι έκανε μάλλον η Γαλλία. Έκανε αυτό το οποίο τη ζητήσαμε να κάνει ακριβώς. Επί τη βάση της οδηγίας του 2004 υπάρχουν τα λεγόμενα διαδικαστικά δικαιώματα ή υλικά δικαιώματα όπως το ονομάζουμε τα οποία υπάρχουν με στόχο την προστασία των πολιτών από απαράδεκτες δράσεις των αρχών, σαν παράδειγμα να συλλαμβάνονται χωρίς λόγο. Αυτά τα διαδικαστικά δικαιώματα δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση του γαλλικού δικαίου και ζητήσαμε από τη Γαλλία ότι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου πρέπει να έχουμε μία απάντηση σε σχέση με το πώς θα αλλάξετε τις νομικές σας ρυθμίσεις εφαρμόζοντας την οδηγία του 2004 για τα διαδικαστικά δικαιώματα και να μας δείξει, ζητήσαμε από τη Γαλλία, ένα αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα σχετικά με την θέση σε ισχύ ε, των ρυθμίσεων αυτών. Λοιπόν, πήραμε την απάντηση αυτή μία ώρα πριν από το τέλος της προθεσμίας. Μία ώρα. Από το Σάββατο το πρωί στις 8 το πρωί εξετάζεται η απάντηση της Γαλλίας προσεκτικά από τους εμπειρογνώμονες και σήμερα νομίζω ότι μπορώ να καταλήξω στο συμπέρασμα ότι όλα τα στοιχεία σε νομικό επίπεδο τα οποία είχε ζητήσει από την Γαλλική Δημοκρατία η Επιτροπή έχουν απαντηθεί. Δεν έχουν όμως βέβαια εφαρμοστεί ε, στο ε, δίκαιο το γαλλικό γιατί πρώτα πρέπει να περάσει από την γερουσία και μετά θα πρέπει να ε, μεταφερθεί de facto στο γαλλικό δίκαιο στις γαλλικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Λοιπόν, εμείς είμαστε ικανοποιημένοι από την απάντηση που μας έδωσαν οι γαλλικές αρχές, αλλά δεν κλείνουμε την υπόθεση. Γιατί έχουμε να κάνουμε με υποσχέσεις, έχουμε να κάνουμε με προτάσεις νομικές οι οποίες δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί. Λέμε λοιπόν ότι εμείς παγώνουμε την δικαστική αυτή διαδικασία αλλά την αφήνουμε φυσικά ανοιχτή μέχρι τη στιγμή κατά την οποία η γαλλική κυβέρνηση de facto στις ε, καθημερινές μορφές εφαρμογής του νόμου αποδεχθεί αυτές τις ρυθμίσεις. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια κάποια νίκη. Για σκεφτείτε τι έχει προηγηθεί μέχρι τώρα. Οι Γάλλοι λένε ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, δεν υπήρχε πρόβλημα, υπήρχε πρόβλημα και τώρα το παραδέχονται και ε, ακριβώς προτείνουν τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Ας δούμε αν θα το κάνουν, εγώ νομίζω ότι θα το κάνουν. Υπάρχει ένα δεύτερο θέμα λοιπόν εδώ. Το δεύτερο θέμα είναι το πώς οι πολίτες κατά τη διάρκεια αυτών των διακοπών του θέρους ε, αντιμετωπίστηκαν, συγκεκριμένοι πολίτες. Ε, είχαν στη δυνατότητά τους σαν Ευρωπαίοι πολίτες σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαδικαστικών δικαιωμάτων τους ή υπέστησαν ε, διακρίσεις. Δεν ξεκινήσαμε εδώ μια διαδικασία επί παραλήψη όπως το κάναμε σε νομικό επίπεδο, γιατί για να μπορέσουμε να δράσουμε μπορούμε να το κάνουμε αυτό επί τη βάση νομικών δεδομένων. Δεν μπορούμε να δράσουμε μόνο και μόνο επειδή μας έχει δημιουργηθεί μια αίσθηση ή ότι είμαστε πεπισμένοι ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα νομικά στοιχεία και γι' αυτό ζητήσαμε λοιπόν από την γαλλική κυβέρνηση να μας δώσει τους φακέλους των μεμονωμένων αυτών πολιτών. Πήραμε αρκετά τους τέτοιους φακέλους. Οι ε, εμπειρογνώμονές μου αναλύουν τους φακέλους αυτούς. Μου είπαν ότι θα έχουν σαφώς συμπληρωματικέ ερωτήσεις να θέσουν προς τη γαλλική κυβέρνηση και πιστεύουν ότι θα τελειώσουν την ανάλυση τους ε, των ερωταπαντήσεων με τη γαλλική κυβέρνηση σε τέσσερις εβδομάδες από τώρα. Λοιπόν αυτές είναι οι δύο θα έλεγα καταστάσεις που ισχύουν μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά. Θα ήθελα να πω με κάθε ειλικρίνεια προς τους ευρωβουλευτές ότι η εφαρμογή της οδηγίας για το 2004 για την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών δεν είναι και ε, πάρα πολύ καλή. Αλλά αυτό το οποίο είδαμε ότι ακριβώς λόγω της επιμονής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι υπόλοιπες χώρες οι οποίες δεν ήταν ε, εξαιρετικές, όχι βέβαια σαν τη Γαλλία αλλά και οι υπόλοιπε χώρε λένε ότι θα εφαρμόσουν τι τις ρυθμίσεις αυτές. Κάτι συνέβη λοιπόν, ε, κατάλαβαν ότι η Ευρώπη δεν αστείευεται και ότι τα δικαιώματα των πολιτών, τα δικαιώματα των πολιτών μας και οι αξίες της κοινωνίας μας είναι σοβαρά πράγματα και θα αντιμετωπιστούν σοβαρά. Αρκετά είπα για την γαλλική περίπτωση έλαβαν τη συγκεκριμένη απόφαση, σας τη μετέφερα, η διαδικασία είναι ανοιχτή. Ας στραφώ τώρα στο θέμα των βάσεων δεδομένων. που πιθανώς περιλαμβάνουν εθνοτικά στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην κατεύθυνση αυτή. Για μια ακόμη φορά πήραμε τη διαβεβαίωση των γαλλικών αρχών ότι όλα είναι σωστά. Εδώ όμως το πλαίσιο είναι διαφορετικό, το σύστημα είναι διαφορετικό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν γαλλικό νόμο για την προστασία των ιδιωτικών δεδομένων και για τη μεταχείριση των ιδιωτικών δεδομένων του οποίου η εφαρμογή ελέγχεται σύμφωνα με τους κανόνες από την ανεξάρτητη αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, το CNIL, Το CNIL λοιπόν πράγματι έχει επιθεωρήσει, έχει ελέγξει και έχει ε, δημοσιεύσει μια έκθεση την προηγούμενη εβδομάδα. Είδατε τα αποτελέσματα της ε, ανεξάρτητης αρχής. Διάβασα και εγώ ε, μερικές φορές ο τρόπος που μεταφέρονται οι επόψεις αυτές των τύπων δεν είναι πλήρης γιατί το ΚΝΙΛ έχει πει πολύ σοβαρά ότι ίσως να μην υπάρχει ε, ανείχνευση εθνοτικών δεδομένων αλλά υπάρχουν επίσης και τράπεζες δεδομένων οι οποίες ε, δεν έχουν υποστεί τον έλεγχο γιατί δεν υπήρξε άδεια από πλευρά των αρμοδίων αρχών. Σχετικά τώρα με τη συμβατότητα των αποφάσεων αυτών με την κοινοτική νομοθεσία, οι πληροφορίες οι οποίες ε, μας έχουν δοθεί έχουν σαν στόχο να καλύψουν τη σωστή εφαρμογή της οδηγίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό αφορά μόνο τις περιπτώσεις που άπονται της μετανάστευσης. Για την μετανάστευση ταυτόχρονα υπάρχει μια σειρά εγγυήσεων και εγγυητικών ρητρών που εφαρμόζονται ονομάζουμε τα δεδομένα αυτά ευαίσθητα δεδομένα και τα ευαίσθητα αυτά δεδομένα μπορούν να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αμφισβητείται το δημόσιο συμφέρον και, και εδώ υπάρχουν ρήτρε ασφαλείας κατάλληλες οι οποίες θα πρέπει ε, να ε, ισχύσουν στη συγκεκριμένη χώρα. Στην περίπτωση που η επεξεργασία δεδομένων δεν καλύπτεται από την Οδηγία Προστασίας των Δεδομένων, τότε η πρόταση απόφαση πλαίσιο μάλλον του 2008 για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση ποινικού δικαίου από πλευράς αστυνομικών και αρχών καταστολής εφαρμόζεται. Σε αυτή την περίπτωση αυτή η οδηγία πλαίσιο εφαρμόζεται μόνον από την 27η Νοεμβρίου του 2010. Επί τη βάση λοιπόν της συγκεκριμένης οδηγίας οι αρμοδιότητες μέχρι τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ιδιαίτερως περιορισμένες. Θα δώσω τώρα και κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις ε, πέραν της γαλλικής περιπτώσεως για άλλες χώρες. Υπάρχουν και άλλες χώρες όπου υπάρχει, υπάρχουν πιθανές τράπεζες δεδομένων που περιλαμβάνουν εθνοτικά ε, δεδομένα ή φυλετικά δεδομένα. Σύμφωνα με την Οδηγία Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, η επεξεργασία τέτοιου είδους ευαίσθητων στοιχείων αδειοδοτείται κατ' και θα πρέπει να γνωστοποιείται στην ε, Εθνική Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Το ΚΝΙΛ πάντα στη Γαλλία στη συγκεκριμένη περίπτωση και οι εξαιρεσει ε, λόγω ακριβώς ε, δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να γνωστοποιούνται και αυτές προς τη συγκεκριμένη επιτροπή. Όταν τέτοιου είδους γνωστοποιήσεις γίνονται η συγκεκριμένη αρχή αυτή είναι σε θέση να αξιολογήσει αν τα μέτρα αυτά είναι συμβατά με τους γενικότερους κανόνες που βρίσκονται σε ισχύ. Και έχω εδώ το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής ανάλυσης την οποία προέβη το ΚΝΙΛ. Και λέγεται εδώ ότι τέτοιου είδους αδειοδοτήσεις δεν ζητήθηκαν από, ε, από αυτό. Ας Προσπαθήσουμε λοιπόν να προχωρήσουμε, να δούμε τι ακριβώς γίνεται από πλευράς των δικαστικών αρχών στη Γαλλία, οι οποίες έχουν την δυνατότητα, σχετίζονται θα έλεγα και είναι υπεύθυνε για αυτού του τύπου τις ενέργειες. Τι γίνεται τώρα στην Ολλανδία. Υπήρξαν αρκετές ε, τράπεζες δεδομένων στις οποίες προεβλέπετο η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και γνωστοποιήθηκαν αυτές προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2005 και το 2006. Τα πιο θα έλεγα προβληματικά στοιχεία αφορούσαν τις ποινικέ δραστηριότητες νέων ε, που προέρχονται από την Καραϊβική ή καραϊβική σε εισαγωγικά καταγωγής. Αυτές οι τράπεζες δεδομένων έχουν καταργηθεί πλέον. Αλλά ένας δήμος στην Ολλανδία θέλει να δημιουργήσει έναν φάκελο εθνοτικών χαρακτηριστικών αλλά ε, θα πρέπει να περάσει μέσα από την Επιτροπή την Ολλανδική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Συνεπώς λοιπόν βλέπουμε ότι οι Εθνικές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι πάντα υπεύθυνε για τέτοιου είδου φακέλους και θα ήθελα να πω προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι εγώ επεξεργάζομαι τη μεταρρύθμιση της οδηγίας προσωπικών δεδομένων με στόχο την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και των δυνατοτήτων παρέμβασης των αρχών προστασίας σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Λοιπόν, ε, προς στιγμήν αυτά είχα να σας πω. Θα πρέπει να διακόψω εδώ, γιατί μετά τα μεσάνυχτα δεν θα έχουμε πλέον διερμηνία, λέει η Επίτροπος. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Θα δώσουμε το λόγο στους ομιλητές εξονομωτός των πολιτικών ομάδων. Δεν διέκοψα την ε, Επίτροπο επειδή έκανε μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση. Θα διακόψω όμω τους συναδέλφους επειδή δεν γίνεται να πάμε μετά τα μεσάνυχτα. Καταρχήν λοιπόν δίνω το λόγο στο Λαϊκό Κόμμα, ομάδα Λαϊκό Κόμμα, τους ματιέ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Ρέντινγκ. Χαίρομαι πολύ που διαπιστώνω ότι σήμερα μας ανακοινώσατε ότι δεν θέλετε να διώξετε την Γαλλία η Επίτροπη. Να θέσω όμως ένα ερώτημα. Πριν κάμπος ο καιρό στην Επιτροπή Λίμπα, σα είχα πει ότι η Γαλλία είχε δώσει όλε τι απαραίτητε πληροφορίε το 2006 και το 2007, όπω επίση και του πίνακες αντισυχία όσον αφορά την μεταφορά των οδηγιών. Τώρα είμαστε στο 2010 και λέτε ότι αυτές οι διαδικαστικές, τα δικαστικά δικαιώματα ε, δεν είναι επαρκή. Δεν μου απαντήσατε λοιπόν τότε όμως κυρία Ρέντινγκ. Όσον αφορά το ίδιο το φάκελο και το μητρό, να σας πω το εξή. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτή τη στιγμή έχουμε πολεμική, αλλά φτάνει πια. Έχετε τα συμπεράσματα της ΚΝΙΛ που η μελέτη της ε, περιλάμβανε προς τον ε, Πρωθυπουργό και εγώ ο ίδιος γνωρίζω πολύ καλά την μελέτη της γαλλικής αστυνομίας, την οποία είχα λάβει και εγώ, κάνατε κάποια πράγματα τα οποία όμως φαίνεται δεν σας βολεύουν. Εσείς ε, θέλετε να προσπιστείτε τα δικαιώματα των μειονοτήτων, όμως θα πρέπει να προσπιστείτε τα δικαιώματα όλων των πολιτών. Να σας πω ότι στη Γαλλία αυτά, αυτά τα μητρώα δεν υπήρξαν ποτέ. Έγιναν έρευνες από την ΚΝΙΛ, κυρία Ρέντινγκ, με ένα συγκεκριμένο αριθμό φοβερών λέξεων κλειδιά όπως ε, τσιγκάνος κλπ. κλπ. και δεν βρήκαν τίποτε από την ΚΝΙΛ, δηλαδή στα αρχεία της γαλλικής αστυνομίας. Το μόνο που θα μπορούσαμε να κατηγορήσουμε την ε, γαλλική αστυνομία είναι, το ότι δεν δήλωσε αυτά, τα, αυτούς τους φακέλους. Οι φάκελοι όμως αυτοί δεν είναι φάκελοι εθνοτικοί ή φιλετικοί. Απλά και μόνο η γαλλική αστυνομία έχει κάποιους φακέλους. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Είμαι η μόνη από το ΕΛΚ, οπότε θα ήθελα να έχω το δικαίωμα να μιλήσω εξωμάτως ομάδος μου. Λοιπόν, αυτοί οι φάκελοι ομαδοποιούν άτομα τα οποία είναι άνευ ε, κατοικίας και δεν έχουν εθνοτικό φιλετικό χαρακτήρα. Εσείς λοιπόν θα μπορούσατε τουλάχιστον να αναγνωρίσετε ότι ναι, ναι, αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Θα πρέπει να το αναγνωρίσετε. Θα ήθελα λοιπόν, κυρία ε, Ρέγντινγκ να σταματήσετε την καχυποψία σας προς την ε, γαλλική κυβέρνηση. Αρχίζει να είναι κακόπιστο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εκ μέρου των σοσιαλιστών ο κύριος Γκυλιόμ για δύο λεπτά. Η ε, κυρία Γκυλιόμ. Επίτροπε, συνάδελφοι, αυτή η πρακτική φιλετική δεν είναι μια νέα πρακτική στι χωρε μέλη, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει εντατικοποιηθεί λόγω ε, τρομοκρατίας, παρανομής μετανάστευσης κτλ. Το γεγονό λοιπόν ότι υπάρχει μητρό για του δρόμου, καταδεικνύει τον επίγοντα χαρακτήρα τη συνέχιση τη έρευνα τη Κομισιόν για αυτό το θέμα, ώστε να διερευνηθεί ακριβώ η νομιμότητα ε, των βάσεων αυτών. Δεν συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό σας κυρία Επίτροπε για την ανακοίνωση της Γαλλία, Χαίρομαι πάντως για αυτά που είπατε. Είπατε ότι η Γαλλία είπε ότι θα μεταφέρει την ελευθερία για την ελεύθερη κυκλοφορία και ότι θα έδινε ένα χρονοδιάγραμμα. Για αυτή λοιπόν την περιβόητη οδηγία και την ένα μεταφορά τη συμβαίνουν τα εξή. Ή λοιπόν ανέλαβε επίσημη δέσμευση η Γαλλία, το οποίο σημαίνει ότι η Κομισιόν δεν έχει λάβει επίσημη απάντηση, ή η Γαλλία έδωσε συγκεκριμένη απάντηση από αυτό το θέμα του και εσεί θα μπορούσατε να είχατε γνώση αυτή τη απάντηση. Επειδή μιλάτε για ένα χρονοδιάγραμμα στην παρέμβασή σα, το χρονοδιάγραμμα αυτή τη στιγμή ισχύει όσον αφορά τη μεταφορά. Αυτή τη στιγμή μεταφέρει η Γαλλία μέσω τη πέμπτη μεταρρύθμιση όσον αφορά τον κώδικα τη μετανάστευση, 7 χρόνια. Εδώ και 7 χρόνια λοιπόν μεταφέρει την οδηγία και να σας διαβεβαιώσω ότι, αυτό πάει πέραν των αρχών των Ευρωπαϊκών για την ελεύθερη κυκλοφορία. Θα πρέπει λοιπόν και εσείς να παρακολουθήσετε για αυτό το θέμα πολύ σοβαρά. Τέλος, ελπίζω να τηρηθεί η αρχή της μη διάκρισης, η Κομισιόν λοιπόν να μην υποχωρήσει και να μην να φοβηθεί τέλο πάντων ή να αξαπατηθεί από τις υποσχέσεις, τις φλούδες της γαλλικής κυβέρνησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εξ ονομάτως της ομάδας Alde Γκρίσμπακ δύο λεπτά. Κύριε Επιτροπή, Πρόεδρε, έστω και αν είναι αργά, η συζήτηση αυτή είναι ένθερμη. Σήμερα το πρωί, μετά από τις σαφείς εξηγήσεις που μας δώσατε, ανακαλύψαμε ένα νέο στο χώρο γαλλικό πληροφοριών ενημερωτικό που μιλούσε για μια παράνομη βάση δεδομένων όπου υπήρχαν τα όνομα, το όνομα το επώνυμο ε, γεωταχή αριθμός κυκλοφορίας όλα αυτά τα στοιχεία τέλο πάντων για αυτούς τους ανθρώπους παρόλο που ταυτόχρονα έλεγαν ότι δεν υπήρχε ένα αντίστοιχο μητρό νομίζω ότι η ύπαρξη του μητρώου αυτού και στις γαλακισάδες χώρες θέτει σοβαρά θέματα διάκρισης. Κυρία Επίτροπε, λοιπόν, τι προτίθεστε να κάνετε και τι άλλα στοιχεία θα έπρεπε να έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιδράσουμε σε σχέση με την παραβίαση της αρχής της μη διάκρισης. Δηλαδή, χωρίς να κάνουμε πολεμικές, να προσπαθήσουμε από κοινού να τηρήσουμε το δίκαιο τόσο στη Γαλλία όσο και στις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες δηλαδή χωρίς πάθη. Οι απελάσεις από την ε, Γαλλία ήταν κάτι το οποίο ήταν αφισβητήσιμο το Μητρό όμως υπάρχει. Με μεγάλο λοιπόν ενδιαφέρον ακούσαμε την ε, συλλογική σας απόψε. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε τι εγγύσει έδωσε στο τέλο τη εβδομάδα η Γαλλία για την τροποποίηση του γαλλικού δικαίου ώστε να μεταφερθεί η οδηγία του 2004. Εμεί λοιπόν και οι συναδελφοί μου θα θέλαμε να συμμεριστούμε την βούλησή σα και την ίδια συλλογιστική ώστε να έχουμε και θα θέλαμε να έχουμε στη διάθεσή μας αυτά τα έγγραφα επειδή είδαμε μετά από την δήλωσή σας απόψε ότι εσείς μάλλον ε, συνθηκολογήσατε για την πολεμική αυτή θα ήταν καλό να ξέρουμε ότι καταρχήν θα πρέπει να πάμε στην ρίζα του προβλήματος θα πρέπει οι ευρωπαϊκές πολιτικές να περισσύνουν των εθνικών πολιτικών όσον αφορά την τήρηση των δικαιωμάτων που αποτελούν τη βάση της ευρωπαϊκής μας δημοκρατίας. Ευχαριστώ για την ομάδα των Πρασίνων, κύριο Δρομεβα για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Όταν εσείς είπατε το περιβόητο enough is enough φτάνει πια πολλοί εδώ στο σώμα αλλά και πολλοί απλοί πολίτες χειροκροτήσαμε. Αυτό δημιούργησε τεράστιες προσδοκίες. Προσδοκίες για όλα εκείνα τα άτομα που ακόμα πιστεύουν, όπως πιστεύουμε εμείς, στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Επιτέλους κάποιος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρθωσε το ανάστημά του και μάλιστα άρθρωσε και τη φωνή του ε, ευδιάκριτα για τα ανθρώπινα θεμελιώδη δικαιώματα που ήταν πάντα στο λάβαρό μας ε, αλλά που πρέπει να τηρούνται στην πρακτική τους εφαρμογή. Μας εξέπληξε κάπως ε, και δεν έγινε από τα κατανοητό όταν ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία η, ότι δεν ελήφθησαν υπόψη ε, τα θέματα της διακριτικής μεταχείρισης αλλά μόνο τα θέματα ελευθερίας της κυκλοφορίας. Αυτό ήταν κάποιο έλλειμμα που υπήρχε. Αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουμε να χειροκροτούμε και να υπερθυμούμε το εγχείρημά σα. Γι' αυτό κάπω δημιουργήθηκε μια σύγχυση σήμερα. Και όχι μόνο για μα, αλλά για όλα εκείνα τα άτομα που προσδοκούσαν και ανέμεναν από τη δική σα δράση να δουν μια γενναία χειρονομία και απάντηση. Και ακόμα περισσότερο σε σχέση με την ε, σχέση που υφίσταται έναντι της γαλλικής κυβερνήσεως ε, που είναι συζητήσιμη η τοποθέτηση της όσον αφορά τη γαλλική κυβέρνηση ιδίως όταν γνωρίζουμε ότι η αναθεώρηση της οδηγίας για την ελευθερία της κυκλοφορίας ε, κινείται μάλιστα σε, κάποιες, σε κάποια πλαίσια που θα έδιναν τη δυνατότητα με μια μεταρρύθμιση πάλι να υποστούν αρνητικές επιπτώσεις και αρνητικές διακριτική μεταχείριση κάποιε ομάδε. Υπό λοιπόν, όλα αυτά δεν θα έπρεπε να υπάρξει συνέχεια και σε αυτή την τάση. Και γι' αυτό σα ζητάμε, σα οικετεύουμε. Παρακαλώ, δώστε μα τη δυνατότητα να έχουμε την ελπίδα όπω την είχαμε σε αυτό το οποίο είπατε. Ότι η ναύφιζη να φτάνει πια και να αρθώσετε το ανάστημά σα έναντι τη γαλλική κυβέρνηση. Αυτό είναι αναγκαίο. Ευχαριστώ. Grazie per il gruppo della sinistra unitaria europea l'onorevole Tavares per un minuto e trenta. Κυρία Επίτροπε, αυτή η συζήτηση είναι για τα θεμελιώδη δικαιώματα, για τη μη αρνητική μεταχείριση και την ελευθερία τη κυκλοφορία. Αλλά έγινε και μια συζήτηση σε σχέση με τις, ε, τη ρύθμιση των εργασιών μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πρέπει να γνωρίζουμε αν ένα κράτο μέλο ε, δρά με καλέ προθέσει σε σχέση με τι πληροφορίε. Και τώρα γίνεται συζήτηση αν εμεί στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είμαστε ικανοί να σεβόμαστε αυτέ τι αρχέ και να είναι αυτέ οι αρχέ σεβαστέ να μιλάμε ειλικρινά και ανοιχτά και να είμαστε σε θέση να είμαστε ανυποχώρητοι στην υπεράσπιση αυτών των δικαιωμάτων. Τώρα για το θέμα των καλών προθέσεων έχουμε απαντήσει σαφεί. Υπάρχουν κράτη-μέλη όπω η Γαλλία που δεν έδρασαν με καλέ προθέσει. Ακόμα και σε σχέση και με τα στοιχεία και τα έγγραφα, σε σχέση με του ε, πολίτε ε, που έχουμε στα χέρια μα. Ακόμα, ακόμα και το καλοκαίρι και υστερότερα. Ε, Έτσι λοιπόν, πώ είναι δυνατόν να λένε ότι δεν υπάρχουν βάσει δεδομένων όταν υπάρχουν υπάρχουν μέσω του ίντερνετ τα στοιχεία αυτά για αυτές τις τράπεζες δεδομένων και ότι υπάρχουν αυτά για τους πολίτες που είναι τσιγκάνοι και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε η σοβαρά υπόψη. Τώρα, στην απάντηση για μια άλλη ερώτηση που είναι και αυτή πολύ σημαντική. Κυρία Επίτροπε, μιλήσατε για μια ιστορική στιγμή και ότι οι ιστορικοί θα κρίνουν για πρώτη φορά αν ήταν σαφή η στάση σα ή όχι. Αλλά υπάρχουν πολλέ αμφιβολίε ε, γι' αυτό, κυρία Επίτροπε. Διότι αμέσω μετά, σε σχέση με την ε, ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΛΥΜΠΕ Πολιτικών Ελευθεριών, υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα στο Financial Times που έλεγαν ότι δεν θα δοθεί συνέχεια σε αυτή την ε, άσκηση προσφυγής επί παραβάση κατά της Γαλλίας ή ότι ήταν συγκυριακή αυτή η δράση. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μπορεί να μιλήσει ανοιχτά και ειλικρινά, τότε θα έχει πραγματικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ω σύμμαχο. Αν διστάσει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα διστάσει να δώσει συνέχεια. Διότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η δράση, όπως είπαμε εμεί εδώ σε τη Βουλή. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Μποργέτσιο απουσιάσει, οπότε δίνουμε το λόγο στους υπόλοιπους ομιλητές. Κόντς για ένα μισή λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κρίση το αίσθημα ασφάλειας των Ευρωπαίων το έχει υπονομεύσει και φυσικά αυτό δημιουργεί και ενδυναμώνει τις ε, ακραίες πολιτικές δυνάμεις. Όμως ε, αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε τέτοια ξεχωριστά φαινόμενα, ότι μια εθνοτική ομάδα ταυτοποιείται και χαρακτηρίζεται κίνδυνος ε, για την κοινωνία ενώ άλλοτε μπορεί να συνδέεται λέει με εγκληματικέ πράξει. Η γαλλική κυβέρνηση συνδέει ε, τους Ρωμά με τέτοιου είδου τράπεζε δεδομένων. Είναι καλό ότι τόνισαν κάποιοι ότι η γαλλική χωροφύλακη εξακολουθεί να συλλέγει τέτοια στοιχεία με βάση την εθνοτική προέλευση πολιτών. Εμεί όμω έχουμε εμπιστοσύνη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω θεματοφύλακα των ε, θεμελιωδών αξιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα δράσει και θα αναλάβει μέτρα δραστήρια κατά τη Γαλλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη αυτά τα στοιχεία για την διατήρηση της δημόσιας τάξης. Όμως είναι απαράδεκτο με βάση την εθνοτική προέλευση πολιτών να συλλέγονται στοιχεία, διότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τα θεμέλια αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης. Οι περισσότεροι Ρωμά ή Τσιγκάν είναι φτωχοί στην Ευρώπη και λόγω της φτώχειας τους πλήττονται από την αρνητική διακριτική μεταχείριση, την μεροληπτική αντιμετώπιση. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι εμείς στην καταπολέμηση αυτής της στόχιας θα έπρεπε να κάνουμε κάτι χειροπιαστά για να είμαστε αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γκρέζ, ένα λεπτό. Σήμερα κυρία Ρέντινγκ μας είπατε με ένα κάποιο ενθουσιασμό ότι η θέση της Γαλλίας δείχνει τη σωστή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν κοινότητα δικαίου και είπατε επίσης ότι θα πρέπει να περιμένουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα επί τη βάση των ευρωπαϊκών αξιών. Έχω εδώ ε, τη συνθήκη και την χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αυτό με κάνει να μην συμφωνώ με αυτά τα οποία είπατε. Τι αποδείξεις θέλετε εσείς. Τι αποδείξεις θέλετε για να καταδικάσετε τις διακρίσεις, ε, τις ε, απελάσεις τις οποίες υφίστανται οι Ρωμά σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Γαλλία. Σίγουρα υπάρχουν μέτρα τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα διαφορετικά ταμεία, αλλά με την στρουθοκαμιλική στάση την οποία υιοθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό υπονομεύεται. Ευχαριστώ. Βερζά, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Ρέντιν και εγώ νιώθω απογοητευμένη σήμερα. Αρκετοί ε, παραδεχθήκαμε τις προηγούμενες δηλώσεις σας, αρκετοί από εμά και σας υποστηρίξαμε. Καταλάβαμε ότι η διαδικασία ε, ε, σχετικά με την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών έχει αναβληθεί η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής Κάθε φορά που σας θέσουμε, σας θέτουμε ερωτήσεις μας απαντάτε με τον ίδιο τρόπο. Και αναρωτιέμαι λοιπόν, σας σέβομαι μένα, αλλά αναρωτιέμαι αν δεν μας κοροϊδεύετε λιγάκι. Ήμουνα στη Μασαλία αυτό το Σαββατοκύριακο και συναντήθηκα με ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται με τους Ρώμ, με τους οποίους εργάζομαι και εγώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχω πραγματικά εντυπωσιαστεί αρνητικά για αυτά τα οποία μου λένε για τους Ρωμά στη Γαλλία. Οι Ρωμά στη Γαλλία έχουν, φοβούνται, κρύβονται, δεν βγαίνουν από τα τροχόσπιτά τους. Τα παιδιά τους δεν τολμούν πια να πάνε στα σχολεία. Δεν μπορούν οι οργανώσεις να τους παρακολουθούν κοινωνικά και σε επίπεδο υγειονομικό. Αυτή είναι η κατάσταση των Ρωμά στη Γαλλία. Αυτά νιώθουν οι Ρωμά στη Γαλλία. Τώρα, ε, για την Τράπεζα Δεδομένων Μέντς. Ας ε, μην εμένουμε εκεί. Η χωροφυλακή δήλωσε ότι το καταργεί. Αλλά ε, για διαβάστε προσεκτικά αυτά τα οποία λέει η ΚΝΙΛ και θα καταλάβετε, Επίτροπε, ότι γίνεται αναφορά στην εθνοτική προέλευση στα πλαίσια των ελέγχων της ΚΝΙΛ Ζητήστε τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. Ζητήστε το σύνολο των ελέγχων τις οποίες έχει κάνει η ΚΝΙΛ. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν έχουμε ε, χρόνο. Θα πρέπει να δώσουμε το λόγο και σε άλλους ομιλητές. Λόμπες Αγουιλάρ, 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επιτρόπε, 9 του Σεπτέμβρη υιοθετήσαμε ένα ψήφισμα που ξεκίνησε μια απαραίτητη συζήτηση. Όλοι αυτοί λοιπόν που θεωρούν ότι οι μετέπειτα δηλώσεις σας ακολουθώντας τις συστάσεις του Κοινοβουλίου και οι εξηγήσει που μας δώσατε από απόψε οδηγούν σε μια απογοήτευση γιατί δεν έχουμε διαδικασία παραβίασης κατά της Γαλλίας και θα πρέπει να επενθυμίσουμε ότι η συζήτηση δεν αφορούσε τη Γαλλία ή ήταν κατά της Γαλλίας, ήταν μια συζήτηση υπέρ των βασικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων, επειδή η Ευρώπη δεν είναι ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και εμπορευμάτων, αλλά κυρίως, κυρίως ελεύθερη κυκλοφορία Ευρωπαίων πολιτών χωρίς διακρίσεις. Βεβαίως και χωρίς φιλετικές διακρίσεις. Αν λοιπόν υπάρχει κάτι το οποίο θα διαρευνήσουμε σε σχέση με αυτά τα μητρώα φιλετικής ε, φύσης, αυτό θα πρέπει να το κάνει η Κομισιόν αλλά η εργασία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί η εργασία αυτή θα πρέπει να λάβει και την επαγρύπνωση, επαγρύπνωση του Κοινοβουλίου ενώπιαν του πειρασμού του λαϊκισμού που αναζητά εξελαστήρια θύματα και όχι απαντήσεις. Αυτή η εργασία λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε, εκτός από να αντιμετωπίσει τον λαϊκισμό και τον πειρασμό του λαϊκισμού, πρέπει να περιλάβει και την δουλειά, σοβαρή δουλειά, για την ενσωμάτωση και ένταξη τον Ρωμά. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια διάσκεψη για την εσωμάτηση των Ρωμά και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να πει ότι αυτή η εργασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Μόλις έχει ξεκινήσει και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας ώστε αν δεν γίνει τελικά η διαδικασία κατά της Γαλλίας να αποδειχτεί ότι αυτή η συζήτηση που έγινε ήταν χρήσιμη και απαραίτητη. Ευχαριστώ. Εντσούγεν Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το 2010 ήταν το ευρωπαϊκό έτος της καταπολέμησης της φτώχειας κατά του κοινωνικού αποκλεισμού. Όμως, εφέτος χάσαμε αυτή τη μάχη. Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όλο και πιο κρίσιμη και δεν βελτιώνονται δυστυχώς τα πράγματα με κανένα τρόπο. Λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν φαινόμενα αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης εις βάρος πολιτών που προωθούνται κιόλας από κυβερνήσεις και βλέπουμε ότι εις βάρος των Ρωμά αυτό έχει ήδη αποδειχθεί ότι υφίσταται ως αρνητική διακριτική μεταχείριση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακας και πρέπει να προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί διαφορετικά θα υπάρξουν κίνδυνοι οι οποίοι θα ελοχεύουν εις βάρος μας. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις αρνητικής διακριτικής μεταχείρισης στα κράτη-μέλη που και αυτές πρέπει να καταπολεμηθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώσει τις ε, διακριβωτικές αυτές ενέργειες και δράσεις και να μην δεχθεί να ασκηθεί πίεση επ' Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ξεκινούμε το Καστέα για ένα λεπτό. Σόγκολ. Σας ευχαριστώ. Η αρνητική διακριτική μεταχείριση με εθνότητα κα αίτια η βάση απαγορεύεται ρητά με βάση το δίκαιο. Παρόλα αυτά υπάρχει όμως η υποψία ότι κάποια κράτη-μέλη ασκούν αυτή την αρνητική διακριτική μεταχείριση εις βάρος πολιτών. Δεν θέλω να μιλήσω για την συγκαλυμμένη όμως αρνητική μεταχείριση, αλλά να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα νομοθέτημα που ανοιχτά και κατάφορα παραβιάζει τα δικαιώματα μιας εθνοτικής μειονότητας. Η νέα σλοβακική κυβέρνηση έχει τροποποιήσει το γλωσσικό νομοθέτημα προς κάποια κατεύθυνση. Παρόλα αυτά όμως επιβάλλονται χρηματικές κυρώσεις ε, πρόστιμα εις βάρος των πολιτών που ομιλούν μια άλλη γλώσσα και ανήκουν σε μια εθνοτική μειονότητα. Βλέπουμε, πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά λοιπόν για αυτή την περίπτωση, ότι αυτό το σλοβακικό νομοθέτημα αβάσιμα την γλωσσική χρήση, την χρήση της γλώσσας της μειονότητας την ε, καταπιέζει. Γι' αυτό ζητούμε από την Επίτροπο όλες αυτές οι πρακτικές και πράξεις ε, να εξεταστούν και όχι μόνο η περίπτωση της Γαλλίας. Ευχαριστώ Μπαντέσκο, ένα λεπτό. Κυρία Επίτροπε, ένα πριν ένα μήνα το Κοινοβούλιο εξέφρασε την ανησυχία του για τη μαζική απέλαση ρωμακής καταγωγής πολιτών. Η Ρουμανία από το 2007 πρόθεσε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ένταξη των Ρώμ που συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβουλίο το Σεπτέμβριο. Υπογραμμίζω ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε καταλήξει καμία ικανοποιητική λύση. Αντίθετα, αυτά που είπαν τα ΜΜΕ σε σχέση με αυτή την βάση δεδομένων στην Γαλλία αφισβητούν την αρχή της μη διάκρισης. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε το γεγονός ότι οι διοικητικές διαδικασίες δεν θα βασίζονται σε φιλετικά κριτήρια. Θα ήθελα εδώ να αποτύσω φόρο τιμής στην δέσμευση τη ε, γαλλική κυβέρνηση για την τήρηση τη ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά την ελευθερή κυκλοφορία. Η Γαλλία και η Ρουμανία θα πρέπει να δράσουν από κοινού ώστε να διευκολύνουν την ε, κοινωνική ένταξη των ΡΟΜ και για την ανέβρεση των ε, απαραίτητων κονδυλίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λούνατσεκ, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η σημερινή συζήτηση καταδεικνύει και πάλι πόσο σημαντική ήταν η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 9 Σεπτεμβρίου ανοιχτά και ξεκάθαρα να πει ότι η Γαλλία, ένα κράτος μέλος, εδώ όπως θεωρούσαμε εμείς, παραβίασε θεμελιώδη δικαιώματα, άσκησε αρνητική διακριτική μεταχείριση εις βάρος πολιτών ε, ε, και στην αρχή σαφέστατα και με κάθετο τρόπο και σαφήνεια απαριθμίσατε όλα αυτά τα οποία κάνατε πράξατε και για τα οποία σας υποστηρίξαμε απόλυτα. Τώρα αυτό το οποίο όμως συνέβη τώρα πραγματικά είναι, όπως πιστεύουμε εμείς, ένα βήμα προς τα πίσω, μια οπισθοδρόμηση το αίτημα δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει μια προσφυγή επί, για παραβίαση της συνθήκης ε, λόγω του ότι εδώ είχαμε στοιχεία το ότι ανήκαν λέει σε μια εθνοτική μειονότητα αυτό αναφέρθηκε ήδη αναφέρθηκε στις ε, ε, γαλλικές ε, εφημερίδες και έχει αποδειχθεί υπήρξε αρνητική διακριτική μεταχείριση βάρος των τσιγκάνων των Ρωμά στη Γαλλία λόγω της ε, εθνοτικής τους αυτής προέλευσης και εδώ και πάλι πρέπει να υπάρξει δραστηριότητα από πλευρά και να να ασκήσετε προσφυγή για αυτόν τον λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. σχέση με αυτή την βάση δεδομένων, να πω ότι αυτές οι βάσεις δεδομένων δημιουργούνται βάσει εθνικής νομοθεσίας και χειρίζονται από εγκεκριμένο προσωπικό. Άκουσαμε λοιπόν, λοιπόν αυτές οι βάσεις δεδομένων στη Γαλλία και στην ε, Ολλανδία και ότι περιλαμβάνουν πληροφορίες σε σχέση με την φιλετική καταγωγή αυτών των ατόμων. Θα πρέπει το θέμα αυτό να διερευνηθεί και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο εδώ υπάρχει παραβίαση των βασικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο, λόγος στον κύριο Σετζένι. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Το κίνημα Ρούμπικ για την Ουγγαρία ξεκίνησε το 2006 και στο στον ποινικό κώδικα η εθνοτική αυτή προέλευση καταγραφόταν και το ότι ανήκε κάποιος ως συγκάνος ε, σε αυτή τη μειονότητα και τα αριστερά μέσα του τύπου ε, αριστερές εφημερίδες ε, παραπονέθηκαν και βλέπουμε ότι χρόνια μετά το ίδιο συμβαίνει και στη Γαλλία και στην Ολλανδία οι τσιγκάνοι θεωρούνται εθνικός κίνδυνος, στοιχείο κινδύνου προσάγονται και σε δικαστήρια επειδή ανήκουν και καταχωρούνται ως εθνοτικοί της τσιγκανικής προέλευσης. Τώρα τι θέλουμε να πούμε. Θέλω να πω στην ε, κυρία από την Σλοβακία που ε, κάχασε και γέλασε για τα θύματα στην Ουγγαρία ότι καταδικάζει την καταχώρηση της, ε, ε, των τσιγκάνων ως εθνοτικής προέλευσης ε, τσιγκανικής και υποστηρίζει όμως το νομοθέτημα για το γλωσσικό θέμα στη Σλοβακία. Ευχαριστώ. Τον, επίτροπο έχει, τον λόγο έχει <laughs> συγγνώμη, επίτροπο Ρέντινγκ. Παρακαλώ να είστε σύντομοι, έχουμε καθυστερήσει πολύ. Πράγματι θα είμαι πολύ συνοπτική. Καταρχάς, ε, δεν, ε, δεν έχουμε καταλήψει τη διαδικασία εις βάρο της Γαλλίας. Έχει υπάρξει μια αναβολή. Περιμένουμε την εφαρμογή των ρυθμίσεων που προτάθηκαν ε, πρακτικά και εμείς δεν θα κρίνουμε τις νομικές προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές είναι, φαίνονται καλές, αλλά πρέπει να εφαρμοστούν. Και τότε μόνο θα κλείσουμε την υπόθεση αυτή. Δεύτερον, για το θέμα των τραπεζών δεδομένων. Το ΚΝΙΛ στη Γαλλία η ανεξάρτητη αρχή ε, κάνει τις επιθεωρήσεις της σύμφωνα με τον γαλλικό νόμο ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι συμβατός με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Και εμείς επαφιέμεθα στις επιθεωρήσεις και στους ελέγχους και την εποπτεία αυτών των αρχών, της ανεξάρτητης μάλλον αρχής γιατί όπως είπα αυτή είναι υπεύθυνη για την ανάλυση και τον έλεγχο. Και νομίζω ότι η ΚΝΙΛ έχει αποδείξει ότι είναι ικανότατη να κάνει τη συγκεκριμένη αυτή δουλειά. Τώρα, αφού τα έχω πει όλα αυτά, νομίζω ότι έχει σημασία σε αυτή τη φάση να επανέλθουμε στην ουσία της κατάστασης πέραν της γαλλικής περιπτώσεως έχουμε 10 εκατομμύρια Ρώμα στην Ευρώπη. Είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μειονότητα. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα η οποία κατοικείται από 500.000 και η Ρωμά είναι 10.000. Ζουν οι Ρωμά στις περισσότερες από τις χώρες μας. Πολλοί από αυτούς σε μια ακραία μορφή ένδυας έχουν προβλήματα κατοικίας, εκπαίδευσης, υγείας, εργασίας και το πρόβλημα δυστυχώς δεν έχει επιληθεί. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό σκάνδαλο, το μεγάλο σκάνδαλο. Ελπίζω λοιπόν ότι ε, τα προβλήματα και οι συζητήσεις ε, θα συνεχιστούν. Θα συνεχιστούν και οι συζητήσεις και αυτό δεν είναι κακό, αλλά αυτές ε, όλες οι κινήσεις θα έχουν σε κάτι βοηθήσει. Να ξυπνήσουν πλέον τα κράτη-μέλη, γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω αυτήν την υπουργική συνάντηση στην Κόρδοβα τον Απρίλιο του 2010, όπου σε 27 χώρες υπήρχαν τρεις οι οποίες εκπροσωπήθηκαν μόνο σε υπουργικό επίπεδο. Λοιπόν, ένα χρόνο μετά θα έχουμε επίσης μια υπουργική συνάντηση Αφού έχουμε κάνει όλη την ανάλυση αυτή με την task force που δημιουργήσαμε για την κατάσταση των Ρωμά και την χρήση ή τη μη χρήση των ευρωπαϊκών πιστώσεων. Θα υπάρξει λοιπόν μια νέα υπουργική διάσκεψη, συνάντηση μάλλον ένα χρόνο μετά, για να μπορέσουμε να δούμε πιο συγκεκριμένα τι προσπάθειες κάνουν τα κράτη-μέλη και ποιες είναι οι εθνικές του στρατιστικές σχετικά με τους Ρωμά. Στα πλαίσια μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής, ενός πλαισίου ευρωπαϊκού. Όλα αυτά φυσικά δεν είναι πάρα πολύ καλά που συμβαίνουν, αλλά έχουν τουλάχιστον βοηθήσει σε κάτι. Τους Ρωμά δεν θα τους παραμερίζουμε πια από εδώ και πέρα, όταν πρόκειται να εφαρμόσουμε συγκεκριμένες πολιτικές για την καταπολέμηση της ακραίας μορφής ένδυας. Αν δεν το πετύχουμε αυτό τώρα που έχουμε την ευκαιρία, δεν θα το πετύχουμε ποτέ. Η επόμενη γενιά των βουλευτών θα εξακολουθεί να συζητά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο αυτά που συζητήσαμε εμείς τις τελευταίες εβδομάδες και αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Ας προχωρήσουμε λοιπόν και ας δράσουμε. Ευχαριστώ ε, κυρία Ρέντινγκ. Η συζήτηση τελείωσε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους υπαλλήλους και την επιμελητία και διαρμηνία για την υπομονή τους.